Ξεκινάμε την συνεδρίασή μας ε, με θέμα την διάδοση φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, Όπως ξέρετε, τα Μη Βασίλειο το... και άλλα, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ, ε, καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν τη διάδοση φορητών όπλων και τον ελαφρύ οπλισμό διότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τομεί όπου είναι γνωστό σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα φορητά όπλα και ο ελευθερή ευλογισμός ξέρουμε ότι προκαλούν του περισσότερου θανάτους τόσο σε εμπόλεμε όσο και σε μη εμπόλεμε περιοχέ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται αυτά τα φορητά όπλα και ο οπλισμός. Επίσης, ε, αυτά τα όπλα μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολλά θύματα ανάμεσα στους πολίτες όσο και σε επίπεδο στρατιωτικό. τα μικρά όπλα και ο ελαφρύ οπλισμός ξέρουμε ότι είναι ευρέως διαδεδομένα και υπάρχει δυνατότητα να αγοραστούν ευκόλως από πολλούς. Κάτι το οποίο διευκρινίζει την ε, διευκολύνει την παράνομη ε, μεταφορά τους. Η περίπτωση τη Λιβύη, όπου ελαφρύ οπλισμός έφτασε στην περιοχή τη Σαχέλ και στα χέρια των ομάδων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη και να γνωρίζουμε ότι αυτά τα όπλα έχουν αποσταθεροποιητική δράση. Αυτή η ακρόαση θα μας βοηθήσει στο να βρούμε τρόπο να καταπολεμήσουμε την διάδοση των φορικών όπλων και του ελαφρύ οπλισμού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε προσκαλέσει τον καθηγητή Κέιφ Κρόουζ, διευθυντή της έρευνας για τα μικρά όπλα στη Γενέβη, ο οποίος θα μας ε, μιλήσει περί αυτών ε, ε, η κυρία Κλάρα Γκάλστραντ, πρόεδρο του Γκόντουν, που θα μας μιλήσει για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να περιορίσει την διάδοση των όπλων αυτών και ο κύριος Μάρκ Μπρόμλε, ο οποίος είναι ερευνητής ό,τι αφορά το πρόγραμμα μεταφοράς όπλων από το Ινστιτούτο της Στοχόλμης και τον κύριο Σέντρικ από το Κέντρο Έρευνας, και Ασφα... Ε, κέντρο Έρευνας και Ασφάλειας. Επίσης έχουμε και ένα άλλο σημείο στην μισά διάταξη. Για το, αυτό το λόγο θα θέλω να δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στον πρώτο μας ομιλητή, τον καθηγητή Κρόουζ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση προκειμένου να σας αναφέρω την ανάλυση μου στο πλαίσιο αυτής της ε, δημόσιας ακρόασης που αφορά στα ελευρά, ελευρό και τα φορητά όπλα. Κοιτάζοντας πίσω ε, μια δεκαετία αναφορικά με το ζήτημα αυτό και ειδικά έχοντας υπόψη την ε, διάσκεψη του ΟΗΕ για, τον, ε, για τα ελαφρά όπλα συμμετέχω σε μια ομάδα ερευνητών που εξετάζουν το ζήτημα της διάδοσης των φορητών όπλων και του οπλισμού. Αυτέ οι απόψει φυσικά που εκφράζω σήμερα εδώ είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Να ξεκινήσω λέγοντα ε, για ποιο λόγο έχουμε τη συζήτηση αυτή σήμερα. Ε, τα όπλα αυτά προκαλούν 526 θανάτους κάθε χρόνο, άμεσα ή έμεσα, ε, τουλάχιστον 40 έως 60% των βίων θανάτων οφείλονται σε ε, ελαφρά όπλα και το 90% εξ αυτών ε, γίνονται σε μη εμπόλεμες περιοχές στην Κεντρική Αμερική, στην Ανατολική και Δυτική Αφρική και σε τμήματα της Αφρικής, της Ασίας, συγγνώμη. Ο ρόλος των ε, μικρών ε, των φορητών όπλων είναι πολύ περιβλόκος και εδώ καλύπτουν μια σειρά από θέματα. Υπάρχει ένας ορισμός του, του ΟΗΕ για τα ε, μικρά όπλα τα οποία περιλαμβάνει ε, τουφέκια, όπλο πυροβόλα, υποπολιβόλα όπως και άλλα όπλα που ονομάζουμε ελαφρύ όπλισμό που πρόκειται για εκτοξευτήρες οβιδών, ρουκετών κλπ. Πριν από 10, χρόνια η εντύπωση που είχαμε για το εμπόριο των φορητών όπλων αφορούσε εμπόρους που τα εμπορευόντουσαν και τα διακινούσαν με πλοία από την Ανατολική Ευρώπη στην, σε περιοχές όπως ε, εμπόλεμη ζώνη της Αφρικής. Καταρχήν να πω ότι υπήρχε μια σταθερή ε, ζήτηση για τα φορητά όπλα και τον ελευθερία οπλισμού. Ε, το, εμπο... το ύψος αυτού του εμπορίου ανέρχεται στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 15% καλύπτεται από τα ελαφρά όπλα και το μεγάλο ποσοστό αφορούσε όπλα όπως τα AK-47, M16, Heckler και Glock, Smith Wesson κλπ. Η παραγωγή μικρών όπλων και ελαφρύ οπλισμού είναι ιδιαίτερα διαδομένο που βασίζεται ε, στις νέε τεχνολογίες. Πάνω από χίλιες εταιρείε σε 98 κράτη ε, εμπλέκονται στην παραγωγή αυτών των όπλων, στα εξαρτήματά τους και η ε, πλειοψηφία αυτών των εταιριών βρίσκονται σε ανεπτυγμένες χώρες. Και όχι μόνο. Φυσικά η παραγωγή αυτών των ε, όπλων δεν περιορίζεται μόνο σε υποπολιβόλα και πυροβόλα, αλλά και σε οβίδες, ρουκέτες κλπ. Η, αύξηση, η ζήτηση όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγαλύτερη σε εμπόλεμες περιοχές όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ κλπ η παραγωγή συγκεντρώνεται στις ε, μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, Ιταλία, Γερμανία, Βραζιλία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο και Ρωσία εξάγουν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Πώς είναι κατανεμμένοι λοιπόν αυτοί οι παραγωγή. Οργανωμένες ε, ένοπλες ομάδες ε, παρουσιάζουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Ένα έως 2% από τα 885 ε, εκατομμύρια φορητών όπλων ανά τον κόσμο. Το 1 τέταρτο χορηγείται στους, στις δυνάμεις και την αστυνομία και ένα χαμηλότερο ποσοστό σε ένοπλες ε, δυνάμεις, σε ένοπλες ομάδες. Λοιπόν, η πρόκληση που βλέπετε σε αυτήν την ε, διαφάνεια δείχνει ότι τα... ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ε, όπλων δεν διαραίουν, δεν διαφεύγουν σε οργανωμένες ε, εγκληματικές ομάδες. Δεν υπάρχουν ε, όμως ε, ικανές αναλύσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, αλλά ξέρουν ότι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό διαφεύγει. Εδώ βλέπουμε τους, τις οδούς που ακολουθεί αυτή η διακίνηση των όπλων. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε την δομή. Έχουμε εδώ τους εμπόρους και βλέπετε παρακάτω πως ε, λειτουργεί η οργάνωση της ε, μεταφοράς και της πώλησης ε, αυτών των ε, όπλων, τα χρηματοδότηση και όπως βλέπω, καταλαβαίνετε και οι σημαίες ευκαιρίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Παρόλο που υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα παράνομα σχετίζονται με διασυνοριακό εμπόριο, ή σε γείτονες χώρες ή παράνομα όπλα τα οποία κυκλοφορούν μέσα στην ίδια τη χώρα από παράνομες ε, ομάδες. Παρόλα αυτά, τα παράνομα όπλα χρησιμοποιούνται στα εγκλήματα και στις σειράξεις. Άρα θα πρέπει να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε πότε τα όπλα περνάνε από τους νόμιμους κατόχους τους ε, παράνομους δηλαδή να μπορούμε να εχνηλατήσουμε την πορεία. Αυτό που ε, έχει σημασία είναι οι διαρροές που μπορεί να γίνουν στην ε, αλυσίδα ε, από αποθήκες, κατά μεταφορές ή από συγκεκριμένες ομάδες διαφθοράς. Στην Αφρική ξέρουμε ότι στις πρόσφατες σειράξεις τα όπλα είχαν εισαχθεί νόμιμα καταρχήν, αλλά στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν με χαμηλή ασφάλεια και γι' αυτό πέσανε στα παράνομα δίκτυα. Επίσης υπάρχει διαρροή και στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολλές ε, χώρες κατέχουν πολύ περισσότερα όπλα από αυτά που χρειάζονται. Μιλάμε για 76 εκατομμύρια, δηλαδή το 1 τρίτον αποτελούν πλεόνασμα πυρομαχικών και γι' αυτό μπαίνουν στα παράνομα δίκτυα. Δεν είναι δαπανηρό να, το να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά χρειάζεται πολιτική θέληση και πολιτικές ασφαλείας. Όπως φαίνεται στη Βόρεια Αφρική μετά από τις πολιτικές αλλαγές στη Λιβύη, εάν δεν υπάρχει έλεγχος, αυτό θα είχε πολλές επιπτώσεις διεθνώς. Σε, σε τις περισσότερες, στις περισσότερες φορές αυτή η διαρροή γίνεται με τη συνενοχή των κυβερνήσεων. Αυτή η διαφάνεια δείχνει ορισμένες από τις πηγές που ε, βρέθηκαν στην κεντροαφρικανική δημοκρατία από αποθήκες σε γείτονες χώρες. Αυτό αφορά το Σουδάν, την Ανατολική Αφρική και χώρες από το κέρας της Αφρικής. Με βάση λοιπόν το παράνομο αυτό δίκτυο, βλέπουμε ότι χρειάζονται παγκόσμια και περιφερειακά επίπεδα. Υπάρχει το, το σχέδιο του 2001 των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ε, πυροβόλων όπλων και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να χνηλατήσουμε την πρόοδο, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή χρειάζεται ένας οδικός χάρτης για να δούμε κατά πόσο ε, μπορούμε να αναχαιτήσουμε την κακή χρήση αυτών των όπλων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν νομικά δεσμευτικά μέτρα όπως ε, το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για τα πολυβόλα του 2001. Φέτος θα έχουμε τις ε, διαπραγματεύσεις για την συνθήκη ανταλλαγής όπλων, εμπορίας όπλων και προβλέπονται και μία σειρά άλλων μέτρων που είναι δεσμευτικά πολλές φορές μέσα στα πλαίσια των περιφερειακών και τοπικών δεδομένων. Εάν τα κράτη εφάρμοζαν όλα τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα δράσης, τότε ο κόσμος θα ήταν ένα ασφαλέστερο μέρος. Επίσης, ως προς την διάδοση των ε, ελαφρών όπλων, βλέπουμε ότι πολλές φορές δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις για να απαλύνουμε αυτό το εμπόριο. Και σε εθνικό επίπεδο χρειάζονται θεσμικές ε, μεταρρυθμίσεις, όπως καλύτερη αυστηνόμευση, ε, καλύτερη ανείχνευση, έλεγχη στα τελωνία, ιδιαίτερα στις χώρες της ε, Αφρικής και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να μην επιτρέπει να επιτρέπει, με συγχωρείτε, την ε, διασυνοριακή συνεργασία. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο νομικό πλαίσιο για να ε, ελέγχουμε την κατοχή και την ε, διάδοση των όπλων, να καταστρέφονται τα πλεονάσματα, να μην συσσωρεύονται δηλαδή και επίσης, τη στιγμή που υπάρχουν κατασχέσεις, να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα. Καλύτερη λοιπόν πολιτική συνεργασία στις εισαγωγές και εξαγωγές. Αυτή η διαφάνεια σας δείχνει και ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση σε σχέση με την πιστοποίηση ως προς τον τελικό χρήστη η παράνομη χρήση όπλων βασίζεται σε παράγοντες ζήτησης περισσότερο και θα πρέπει να δούμε πώς θα ελέγξουμε αυτό το δίκτυο ζήτησης. Θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας και ε, μειώσεις της ε, χρήσης τα Ηνωμένα Έθνη δεν έφτασαν σε μια συμφωνία στη διεθνή τους διάσκεψη, όμως το 2012 η κατάσταση είναι διαφορετική, γιατί βλέπουμε ότι τα, ε, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο μπόρεσαν να εφαρμόσουν ήδη υπάρχουσες συμφωνίες. Σε έναν ιδεατό κόσμο θα υπήρχαν θεσμικά δεσμευτικές συμβάσεις. Στον πραγματικό κόσμο όμως θα πρέπει να προτείνουμε ορισμένους ε, στόχους. Καταρχήν να ορίσουμε έναν επίσημο μηχανισμό για την αποτίμηση προόδου και εφαρμογής της δράσης των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, να μπορέσουμε να ορίσουμε καλύτερα τρόπους αρρωγής να θέσουμε ένα τυπικό πλαίσιο για τη διαδικασία παροχής ε, διεθνούς συνεργασίας και αρρωγής και να συμφωνήσουμε στις διαπραγματεύσεις για διεθνή μέσα έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως προς τους μεσάζοντες και την πιστοποίηση ως προς τους τελικούς χρήστες. Επίσης να ενισχύσουμε το διεθνές μέσον ιχνηλάτησης, ιδιαίτερα για ένα μηχανισμό αρρωγής και τελικής ιχνηλάτησης. Επίσης, θα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχη και συναντήσεις μεταξύ κρατών. Νομίζω ότι η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με την ε, χρήση από μεμονωμένους, δηλαδή ε, χρήση όχι στρατιωτική αλλά πολιτική. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μία ε, συμμετοχή, ευρύτερη μετοχή, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι τα όπλα αποτελούν ένα στοιχείο μέσα στα πλαίσια του διεθνούς εγκλήματος και αυτό που έχει σημασία είναι να κρατήσουμε να υπάρχει ε, δημόσια ασφάλεια. Γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε όχι μόνο με τον ε, έλεγχο των όπλων, αλλά και την απονομή δικαιοσύνης παγκοσμίως και εθνικός. Πιστεύω ότι υπάρχει ευρύ φάσμα για δράσεων για να μπορέσουμε να μειώσουμε την ε, χρήση των μικρών ελαφρών όπλων και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα είδος αφοπλισμού καθώς και προγράμματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των όπλων. Αυτό είναι μόνο ένα από τα θέματα. Πολλά μπορούν να γίνουν έμπρακτα και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ε, ηγετικό ρόλο. Σας έδωσα μόνο μία μερική εικόνα, ελπίζω όμως να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε κατά τη συζήτησή μας. Now, Mrs. Clara Gansland. Κυρία Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ σήμερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν στην ε, μείωση της ε, προωθήσεως των μικρών όπλων ε, σχετικά με, την, με τα θέματα των μικρών όπλων είμαι υπεύθυνη για την εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση του προγράμματος για την καταπολέμηση της παράνομης διαδόσεως των απλών όπλων, ε, οπλισμών και ε, των ε, την πάταξή του. Ασχολούμαστε με την νόμιμη μεταφορά των μικρών όπλων και ε, τις σχετικές δραστηριότητες. Ε, υπάρχουν ε, ε, ε, ε, υπάρχει λοιπόν ένα θέμα στο οποίο εγώ θα επικεντρωθώ, δηλαδή την παράνομη διάδοση των όπλων αυτών και όσον αφορά την, το νόμιμο εμπόριο αναφέρομαι στον κύριο Ντελαπιάτσα ο, ο οποίος στη συνέχεια θα παρουσιάσει το θέμα αυτό. Οπότε από το 2001 έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα επίποδα περιφερειακά και σχετικά με συγκεκριμένες χώρες για να καταργήσουμε το παράνομο εμπόριο μικρών όπλων και αυτό συμπληρώνει το πρόγραμμα δράσεως το οποίο είχε θεσπιστεί το 2005 για να καταπολεμήσουμε τη διάδοση των μικρών όπλων ε, και ε, των σχετικών ε, δράσεων Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και γι' αυτό θα αναφερθώ καταρχήν στο πρόγραμμα δράσης που θα οργανωθεί εφέτος το καλοκαίρι διότι μας δίδεται μία πολύ καλή ευκαιρία όχι μόνο να επαναλάβουμε την ανάγκη να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης και να προωθήσουμε την εξάπλωση του προγράμματος αυτό αλλά και να την ενισχύσουμε. Δεδομένων των συνεδριάσεων που είχαμε φέτος πλησεύουμε ότι η συνεδρίαση αναθεώρησης θα πρέπει ε, να δει πώς μπορούν τα ισχύοντα προγράμματα να λιλοενισχυθούν ε, αμοιβαία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής έχει συμμετάσχει σε όλες τις συζητήσεις και υποβάλλει έγγραφα εργασίας για αυτή την αναθεωρητική διάσκεψη τις οποίες μπορεί καλής να συμβουλευτεί στο διαδίκτυο. Έχουν υπάρξει ε, συζητήσεις για τα προγράμματα αυτά και παρόλο που διαφέρουν οι γνώμες, ιδίω όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για μη κρατικούς συμμετέχοντες, οι αποφάσεις που χρειάζονται για την αναθεώρηση και την προετοιμασία θα πρέπει να προχωρήσουν βάσει της ε, ε, σύνοψης την οποία ε, και των πορισμάτων που παρουσίασε η Προεδρία της Νικηρίας. Πέραν αυτού όμως θέλουμε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα αυτό και γι' αυτό σας ενθαρρύνω να εξετάσετε όλο το έγγραφο το οποίο όπως σας είπα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τις συστάσεις μας θα ήθελα να τονίσω καταρχήν την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για να διαχειριστούμε τα αποθέματα, να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά τους και την καταστροφή τους. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ε, των τελωνιακών αρχών που να ενισχυθούν και των νομικών αρχών όπως και των δικαστικών για να μειωθεί η διακίνηση διασυνοριακά αυτών των οπλισμών. Χρειάζονται ε, μηχανισμοί που πρέπει να αναπτυχθούν σε διάφορα επίπεδα για να να υπάρχει ε, μεγαλύτερη δυνατότητα αδειοδοτήσεων και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα εμπάργο διακινήσεως όπλων. Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες και τις ειρηνευτικές αποστολές θα πρέπει να βασίζονται σε ανταλλαγή πληροφοριών και ειρηνευτικές ε, δράσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν ε, την ασφαλή αποθήκευση και την ε, καταστροφή των, οπλισμών, των μικρών οπλισμών και να παρακολουθούνται και από την Ίντερπολ ε, και από ένα ενιαίο σύστημα παρακολουθήσεως των κλεμμένων ή χαμένων τέτοιων οπλισμών. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να πείσει τα κράτη-μέλη ότι αυτά τα βασικά βήματα είναι σημαντικά για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και την καταπολέμηση της διαδόσεως των ε, όπλων αυτών που θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα που αναφέρονται αναφέρονται στη στρατηγική. Ε, απλώς ε, θέλω να αναφερθώ στις ε, τεράστιες ποσότητες τέτοιων αποθεμάτων στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι σχετικές δραστηριότητες που έχουν παρακολουθήσει από την αρμόδια υπηρεσία την ΣΥΣΑΚ στη, στα Ανατολικά Βαλκάνια θεσπίστηκε το 2010 για ασταθή αποθέματα εξοπλισμών και πυρομαχικών. Ε, στα πλαίσια αυτά Έχω ε, υπάρξει ανάπτυξη στα Ανατολικά Βαλκάνια ενός συστήματος καταγραφής και μετά την λήψη της αποφάσεως του Συμβουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί στενά με τις εμπλεκόμενες χώρες για να βοηθήσει ε, την διαχείριση των αποθεμάτων αυτών των όπλων, την καταγραφή τους και την καταστροφή τους για να αποφύγει να διανεμηθούν περαιτέρω. Δεύτερον, για να εφαρμοστεί το εμπάργο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει την απόφαση η οποία θα απαγορεύει ε, την ε, διακίνηση αεροπορικός αυτών των ε, όπλων που εξασφαλίζεται σήμερα από τον Σύπρη που εκπροσωπείται εδώ σήμερα και θα πρέπει ε, να παρακολουθούνται τα ύποπτα αεροπλάνα τα οποία ενδέχεται να, είναι, να έχουν εμπλακεί σε τέτοια διακίνηση. Έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα και γνωρίζουμε τις εταιρείε και τα αεροπλάνα τα οποία εμπλέκονται στην διακίνηση αεροπορικός των μικρών όπλων και οπλισμών. Επιπλέον έχει ληφθεί μία απόφαση του Συμβουλίου η οποία συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Αφοπλισμού και που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεως των εκπαιδευτών στη Δυτική Αφρική, την κατάρτιση εγκαταστάσεων σε χώρες όπου δεν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις στήριξη της συμπλήρωσης και εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών για, την, ε, ε, ε, για τους οπλισμούς αυτούς στην περιοχή των μεγάλων λιμνών στην Αμερική όπως και στη Λατινική Αμερική και Πλέον αυτού, το κατόψη αποφάσεως του Συμβουλίου, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά στο ε, στην κατάρτιση ενός πλαισίου σταθερότητος και αυτό το πλαίσιο στηρίζει την Interpol για να αναπτυχθεί μία βάση δεδομένων σχετικά με τα κλαπέντα όπλα και ε, όλα τα στοιχεία δίδονται στην Ίντερπολ για να μπορεί να παρακολουθήσει τις κινήσεις των όπλων αυτών μέσω των συστημάτων της. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάζει και φροντίζει να έχει μία σταθερή ρήτρα κατά της εξαπλώσεως αυτών των παρανόμων οπλισμών σε όλες τις συμφωνίες της για να αντιταχθεί στις συσσόρευση παρανόμων τέτοιων όπλων διεθνώς. Και τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο προωθεί την ε, ε, κατάργηση ε, αυτών των οπλισμών αλλά και στον πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες το επαναλαμβάνει και τώρα ετοιμάζουμε ένα νέο σχέδιο αποφάσεως του Συμβουλίου για να περιορίσουμε την τον κίνδυνο παρά, ε, παράνομης διακίνησης μικρών όπλων εις τον χώρο του ΟΑΣΕ. Ε, και έχοντας υπόψη την κατάσταση στο Κυργιστάν και στη Λευκορωσία ε, και την συσσόρευση όπλων σε αυτές τις περιοχές ζητούμε να υπάρξουν εφαρμογές που θα παρακολουθούν τα όπλα αυτά σε πολλά κράτη του ε, ΟΑΣΕ Τέλος, ε, όσον αφορά το πρόγραμμα ελέγχου μικρών όπλων ή στην Αμερική, θα συμβάλλει εις ε, την, ε, τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης αυτών των όπλων στην Κεντρική και Νότιο Αμερική. Και είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί σειρά θανάτων καθημερινά και όλες οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις οι οποίες ε, υπάρχουν απειλούν την ε, ειρήνη εξού και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει ε, την, την παρακολούθηση αυτών των όπλων διεθνών και να βοηθήσει τα κράτη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο να ελέγχουν αυτού αυτούς τους οπλισμούς και να, μίλη να μειώσουν την ένοπλη βία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρκ Μπρόμλεϊ από το Διεθνές το Ειρήνη στη Στοχόλμη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το, το σημαντικό ζήτημα το οποίο το 2012 έχει αποφύσει τα φώτα της δημοσιότητας μετά από τα όσα συμβαίνουν στον ΟΗΕ και στην ΟΝΟΣΑ. Ε, Σε μια σύντομη παρουσίαση δεν μπορώ φυσικά να εξετάσω όλες τις πτυχές του ζητήματος. Ε, μου είπαν να μιλήσω για προτάσεις σχετικά με τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης. Θα μιλήσω για ζητήματα που αφορούν την αποθήκευση και την διαχείριση των ε, αποθεμάτων, κάτι το οποίο εξετάζεται αυτή την περίοδο. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπες, τρόπους για την διάδοση των φορητών όπλων και του ελευθερού οπλισμού. Χαίρομαι που οι δύο προραλήσαντες έδειξαν αυτά τα αισθήματα. Θα ήθελα τώρα να σύντομη παρουσίασή μου να μιλήσω για τον έλεγχο της μεταφοράς όπλων ειδικά σε ό,τι φορά τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό, που είναι ο βασικός τομέας με τον οποίο ασχολείται το ΣΥΠΡΙ. Τα κράτη-μέλη έχουν ασχοληθεί ενεργά με το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να σας αναφέρω τώρα πού μπορούν να, να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε ό,τι αφορά την αποθήκευση και τη διαχείριση των αποθευμάτων. προκειμένου να περιορίσουμε και την ε, παράνομη μετακίνηση, διακίνηση αυτών των όπλων και του ελεύθερου όπλισμού ανά τον κόσμο. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τρεις τομείς που αφορούν στην μεταφορά φορητών όπλων και που έχουν άμεση επίπτωση στην διάδοση αυτών έχουν συμπεριληφθεί στην στρατηγική μας το 2005 και υπάρχουν τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης υπάρχουν τομείς όπου υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν περαιτέρω προσπάθειες. Τώρα θα αναφερθώ πρώτα στον έλεγχο και την δίωξη των μεσητών φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, να επιβληθεί ένα εμπάργκο των ΗΕ και την ε, ε, συνεργασία που μπορεί να υπάρξει στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την μεταφορά αυτών. Τώρα το, πρώτο ζήτημα, όπως είπαμε, τον έλεγχο των ε, μεσαζόντων, όταν φτάσουμε τη δεκαετία του 1990-2000, υπήρχαν πολλέ προτάσεις από κυβερνήσεις και από φορείς ε, του ΟΗΕ για την προσπάθεια περιορισμού αυτής της διακίνησης ε, ε, μην ξεχνάμε την περίπτωση της Ρουάντα, της Αγγόλα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, την Λιβερία και την Σιέρα Λεόν για κατά την περίοδο των ε, των σειράξεων. Έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από νομικά δεσμευτικά μέσα τα οποία προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ελέγχου, ειδικά η κοινή θέση του Συμβουλίου του 2003 θέτει τα ελάχιστα πρότυπα για ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να φάρουν τα κράτη-μέλη για τον έλεγχο της εμπορίας, του εμπορίου. Υπήρξε μια σημαντική ε, επέκταση της εντολής και της δυνατότητας ε, δίωξης εταιριών αλλά και προσώπων που εμπλέκονται σε αυτήν την διακίνηση. Αλλά θεωρώ ότι εδώ υπάρχουν κάποια κενά, ιδιαίτερα στον τομέα της εφαρμογής. Προφανώς ε, έξι κρατημένοι ε, εφάρμοσαν απόλυτα την συμφωνία αυτή 10 χρόνια μετά από την συναψή της βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια παραδείγματα για το πώς τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν και παραβίασαν αυτήν την συμφωνία. Το ζήτημα της δίωξης προσώπων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε αυτήν την διακίνηση είναι κάτι το οποίο φροντίσαμε να προωθήσουμε τον τελευταίο καιρό και ήδη έχουμε πετύχει την δίωξη πολλών ε, εμπλεκομένων ε, το Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο θέλει να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες και τις εξουσίες που έχει για να διώκει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διακίνηση όπλων και πυρομαχικών. Βλέπουμε ότι από πλευρά κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέλουν, υπάρχει βούληση για την ε, εφαρμογή της ε, νομοθεσίας αυτής. Τα τελευταία χρόνια είχαμε την κυβέρνηση του Βασιλείου, το οποίο ξεκίνησε δύο σημαντικές διώξεις, αλλά και παραδείγματα, άλλα, άλλα παραδείγματα είναι δύσκολο να εντοπίσουμε και να βρούμε Τα κρατημέλη θα πρέπει λοιπόν να εντείνουν τους ελέγχους τους σε ό,τι φορά τη διάδοση φορητών όπλων και ελεύθερων όπλισμού και να εξετάσουν ε, τις, ε, τις πρακτικές που εφαρμόζονται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, έλεγχος και δίωξη και σε εθνικό επίπεδο. σε ορισμένες περιπτώσεις ε, η έλλειψη εμπειρίας ε, για το πώς μπορούν να ασκηθούν αυτές οι διώξεις ε, οδηγούν σε περίπλοκες υποθέσεις. Σίγουρα θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για το πώς θα πρέπει να δρουν τα κράτη και σε διεθνές επίπεδο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και την εξέταση αποτελεσματικών ε, περιπτώσεων στις οποίες ε, η δίωξη ε, κατέληξε σε αίσιο αποτέλεσμα. Περνώντας τώρα στο δεύτερο ζήτημα, την επιβολή του εμπάργου στρατηγική της Ευρωπαϊκής για τα φορητά όπλα και δηλαδή από το 2000, 2000 ήταν να ε, προωθήσει τις κυρώσεις αλλά και την ε, εποπτεία. Ε, Πρόθεσε την ανταλλαγή προφοριών ιδιαίτερα σε ό,τι φορά την παρακολούθηση της εφαρμογής και υλοποίησης του εμπάργου του ΟΗΕ. Και για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου που αφορούσε την έλεγχο διάερος Φυσικά θα πρέπει να χορηγούνται στοιχεία στις ε, τελωνιακές αρχές. Νομίζω ότι η σύπρι που δουλεύει πάνω σε αυτό το ζήτημα είχε αποτελέσματα ιδιαίτερα καρπο, αποδοτικά. Υπάρχουν ε, ομάδες εμπειρογνώμων του ΟΗΕ, τις οποίες ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, και ασχολείται με τις ε, παραβιάσεις. Αυτά τα, αυτές οι ομάδες τα τελευταία χρόνια έτυχαν χαμηλής χρηματοδότησης, δηλαδή χαμηλότητας από το παρελθόν. Οι ομάδες αυτές των εμπειρογνωμόνων ε, πρόσφατα ήταν ε, η βασική πηγή πληροφοριών αλλά δυστυχώς το τελευταίο καιρό είδαμε ότι έγιναν σημαντικές περικοπές ε, στη χρηματοδότηση και αυτό σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται σε πολιτικές πιέσεις που ασκήθηκαν. Τώρα, ε, πώς μπορεί να αναμειχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το ζήτημα. Με, σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συστήσει τους δικούς της, ε, δικές της ομάδες εμπειρογνωμόνων. Ε, έχουμε φυσικά τους εμπειρογνώμονες από πλευράς ΟΗΕ που ασχολούνται με το θέμα αυτό, αλλά έχουμε και εμπάργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουμε όμως το απαραίτητα τους απαραίτητους φορείς, τους απαραίτητες ομάδες για να ασχοληθούμε με την εφαρμογή αυτού του εμπάργου. Ε, δεν θέλω να πω εδώ ότι πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση ή κάποια δικαστική οργάνωση που να ασχοληθεί με αυτό. Όπως και τα, οι ομάδες του ΟΗΕ θα πρέπει να εξετάζουν τις περιπτώσεις παραβίασης του εμπάργου ή και την συμμετοχή κάποιων οργανώσεων ή επιχειρήσεων. Αυτέ οι προφορίε λοιπόν θα διευκολύνουν τον διάλογο, θα δουν ε, κατά πόσον εφαρμόζεται ορθά το εμπάργκο και αυτό φυσικά τα αποτέλεσμα θα πρέπει να δίνονται και στους οργανισμούς ε, αδειοδότησης Τώρα για την εφαρμογή του εμπάργου, ένα το τομέες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει δράση είναι κατά πόσο πρέπει να υπάρχει μια λεπτομερής αξιολόγηση για το πώς ε, εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις τους ε, τόσο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυτές, αυτά τα εμπάρκο, είναι οι αποκλεισμοί επιβάλλουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τις ε, διατάξεις ε, και σε επίπεδο εθνικό αλλά και σε διεθνές. Πρόσφατα είδαμε περιπτώσεις όπου η έλεγχη, αυτού του είδους έλεγχη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη. Εντάξει, υπάρχει μια έλλειψη σαφήνειας, ακρίβειας αναφορικά με το ποιε είναι οι αρμοδιότητες των κρατών. Ίσως λοιπόν εδώ να αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι αποφάσεις ε, του ΟΗΕ αναφορικά με το εμπάργο. Και κάτι ακόμα που αφορά στους ελέγχους. Ε, φτάνω στο, πάλι στο 2005 στη στρατηγική που αποφασίσαμε για την κατάσταση που ακολουθούσε στην Αφρική Χρειάζεται λοιπόν να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε τα κράτη της περιοχής. Έχουν γίνει πολλά, δεν ε, το αμφισβητεί κανείς. Η βοήθειά μας, η αρρωγή μας λοιπόν προς αυτές τις περιοχές είναι απαραίτητο να συνεχιστεί. Και τέλος, τροφή προσκέψη, εάν ε, πάμε πίσω στην, διάδοση, στην Ισραηλική για τη διάδοση φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, πέραν του ότι θα πρέπει να υπάρχει συνδρομή για τον έλεγχο αυτών, αλλά θα πρέπει να προάγουμε και τον έλεγχο στα στις βιομηχανίες που παράγουν αυτά τα όπλα. Θα δούμε επίσης πώς μπορούμε να μετατρέψουμε στρατιωτικές ε, εγκαταστάσεις ε, σε οι οποίες εξάγουν ε, παρόμοια όπλα Το όλο ζήτημα λοιπόν της μετατροπής που συζητήθηκε μετά από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις ε, συνεχίζουν να λειτουργούν και να παράγουν ε, φορητά όπλα και ελαφρύ οπλισμό με χαμηλό κόστος. Και το αποτέλεσμα είναι η ε, αποσταθεροποίηση περιοχών. Ίσως θα πρέπει να, να επανεξεταστεί το ζήτημα της ε, μετατροπής που είχε ξεκινήσει το 2005 και αυτά σε εγκαταστάσεις, αυτές μηχανίες ε, να ε, μετατραπούν και να παράγουν άλλα προϊόντα. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Πέρκιν από την Κομισιόν, την Επιτροπή Ασφάλειας, Ασφάλειας. Θα ήθελα να μιλήσω στα γαλλικά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πρώτες περιφερειακές οργανώσεις που θεώρησε ότι η διάδοση των όπλων και των πυρομαχικών είχε σημασία για την ασφάλεια και την ανάπτυξη των περιφερειών του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να καταπολεμήσει την συσσόρευση και την διάδοση των όπλων. Άρα το 2005 ενέκρινε μια στρατηγική για να διαρθρώσει αυτές τις πράξεις σε ένα συνολικό πρόγραμμα δράσης για να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στην πολιτική ασφάλειας και ανάπτυξης. Αυτή η δράση βασίζεται σε δύο άξονες. Καταρχήν, η προώθηση της πολυμέρειας με την ενίσχυση μέσων και κανονισμών σε διεθνές επίπεδο, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, και προωθεί και αυτή τη δράση στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, ως δεύτερη δράση, βρισκόμαστε στις χώρες και στις περιφέρειες που έχουν πληγεί, όπου γίνεται διάδοση των ελαφρών όπλων με τη δραστηριότητα και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Δύο δράσεις ορίστηκαν το 2005 υπό Σαχάρια Αφρική όπου θεωρείται ότι είναι ο πιο αποσταθεροποιητικός παράγων διάδοσης ε, ελαφρών όπλων και η Ανατολική Ευρώπη για το ρόλο που έπαιξε στη διάδοση των όπλων, ιδιαίτερα στην Αφρική. Άρα προσπαθούμε να δράσουμε και προληπτικά αλλά και αντιδρώντας τις υπάρχουσες καταστάσεις. Το φάσμα δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά τις Βρυξέλλες βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της διάδοσης των ελαφρών όπλων. Γιατί τονίζουμε ότι με βάση τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, RSS, και με την ενίσχυση άλλων οργανώσεων, καταπολέμησης της διάδοσης των ε, ελαφρών όπλων προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτή τη διάδοση στην υποσαχάριο Αφρική και στην Ανατολική Ευρώπη. Όμως δεν θίγουμε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τη διάδοση των όπλων. Η δράση βασίζεται μόνο στην παράνομη διάδοση ορίζοντας ένα, ε, μία γραμμή διαχωρισμού ανάμεσα στη διάδοση, στην παράνομη διάδοση ή στη διάδοση γενικότερα. Όμως υπάρχει και υπάρχουν και τα όπλα που κατασκευάζονται νόμιμα και διαδίδονται νόμιμα. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε τους κανονισμούς τη στιγμή που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Όταν μιλάμε για την παράνομη διάδοση θα πρέπει να δούμε ποια, ποιο είναι το μέρος της δραστηριότητας το οποίο είναι νόμιμο και μετά μετατρέπεται σε παράνομο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι με βάση τις πολυμερείς σχέσεις θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να προωθήσουν τη διάδοση αυτή έτσι ώστε εξάγοντας να ελέγχουν τις εξαγωγές. Γιατί δεν ξέρουμε, ε, ξέρουμε με συγχωρείτε, ότι εξάγουμε και μιλάμε για ένα ύψος δαπανών και εσόδων της τάξης των δύο δις. Δύο πρωτοβουλίες έχουν αναλυφθεί. Η πρώτη αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών και η δεύτερη την μεσητεία. Βασιζόμαστε λοιπόν στη δυνατότητα των κρατών μελών να θέσουν σε εφαρμογή αυτή την ομοθέσια σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η έλλειψη συντονισμού και ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εξαγωγών όπλων περιορίζουν την εναρμόνιση αυτών των πολιτικών ιδιαίτερα σε σχέση με την στρατηγική καταπολέμηση της διάδοσης ελαφρών όπλων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για χώρες που ευεργετούνται από προγράμματα αρρωγής μέσα στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής. Γιατί τα ελαφρά όπλα μεταφέρονται σε όμορες χώρες από τις χώρες επέμβασης που έχουν υψηλά αποθέματα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην παράνομη διακίνησή τους. Το παράδειγμα της Λιβύης μιλάει από μόνο του. Το ίδιο αφορά τον αποκλεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε ο Μαρκ Μπρόμλι, γιατί τα 27 κράτη-μέλη προβαίνουν σε μία απόφαση, λαμβάνουν μία απόφαση, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τη θέσουν σε εφαρμογή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση του ρωσικού πλοίου που οι αρχές της Κύπρου άφησαν να μεταβεί προς τη Συρία με τα πυρομαχικά που μετέφερε. Προσπαθούμε να δράσουμε μέσα στα πλαίσια προτεραιοτήτων που μπορούν να αναλυφθούν στα πλαίσια της στρατηγικής όπως προϋπάρχει και στα πλαίσια της μεταφοράς ελαφρών όπλων. Όσον αφορά την στρατηγική, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τις πολυμερείς σχέσεις και υπ' αυτή την έννοια η 27 στην διάσκεψη και διαπραγματεύσεις της συνθήκης για την εμπορία των όπλων, οι 27 θα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά πώς θα ε, δράσουν μέσα στα πλαίσια των ε, ελαφρών όπλων. Ως προς την αρρωγή, θα ήθελα να μιλήσω για τη διαχείριση των αποθεμάτων ελαφρών όπλων και των ε, σχετικών πυραμαχικών και στην καταστροφή τους. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την διάδοση των ελαφρών όπλων, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και ακόμα κι αν είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τη δραστηριότητα βράχη και μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη δράση της γενικότερα μετά από 10 χρόνια ευρωπαϊκής και διεθνούς αρρωγής για την καταπολέμηση της διάδοσης των ελαφρών όπλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλύσει τα μέχρι τώρα πεπραγμένα. Και άρα η έγκριση μιας συνθήκης για το εμπόριο των όπλων θα βοηθήσει σε, στο άνοιγμα ενός νέου κύκλου αρρωγής και συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Η Ένωση θα πρέπει να ξαναδεί τη στρατηγική στο σύνολό της. Οι παρεμβάσεις, οι επεμβάσεις είναι αρκετές. Ποιες είναι οι κατά προτεραιότητα ζώνες όπου θα πρέπει να δράσει η Ένωση. Πώς οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να συντονιστούν με τις μεμονωμένες ε, πρωτοβουλίες των κρατών μελών και πώς μπορεί να ορίσει καλύτερα τη στρατηγική της με βάση τις εξαγωγές των κρατών μελών. Την παρούσα στιγμή υπάρχει μια συλλογική απόφαση, της, ε, η, η λήψη μια συλλογικής απόφασης ε, δεν φαίνεται εφικτή, όμως μπορεί κανείς να δράσει τουλάχιστον ε, άναντι θα πρέπει να απαιτήσουμε από τις χώρες εισαγωγής ελαφρών όπλων να ορίζουν, να δεχτούν μία ρήτρα η οποία ε, ονομάζεται New for Old που απέτησε η Γερμανία ήδη από το 2003 για να αποκλείσει την, ε, το πολλαπλησιασμό της διάδοσης αυτών των όπλων. Και εάν λάβουμε υπόψη το η βαρύτητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην ε, αγορά ελαφρών όπλων, θα ήταν ε, πολύ δύσκολο για έναν εισαγωγέα να αρνηθεί τη ρήτρα αυτή και να αναζητήσει όπλα αλλού. Ένας καλύτερος συντονισμός των εξαγωγών της Ευρώπης θα μπορούσε να γίνει με την ε, ενημέρωση ενός καταλόγου των στοχοθετημένων χωρών μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής και να μην επιτρέψουμε την επανεξαγωγή προς αυτές τις χώρες. Έτσι θα μπορούσαμε να αναχαιτήσουμε τη διάδοση ελαφρών όπλων προς αυτές τις χώρες. Παράλληλα θα πρέπει οι 27 να ορίσουν πού γίνονται, πού υπάρχουν διαρροές και διαφυγή έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να προβεί σε μία πλήρη ανάλυση του κινδύνου, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της διάδοσης. Έτσι θα επιτύχουμε και μία μεγαλύτερη εναρμόνιση. Θα πρέπει να υπάρχει εποπτικός μηχανισμός στην περίπτωση εμπάργο και θα πρέπει να υποστηρίξει το πάνελ εμπειρογνωμόνων μέσα στα πλαίσια των εμπάργων που ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, τη στιγμή που αμφισβητούνται από ορισμένα κράτη. Άρα οι χώρες υπό αποκλεισμό είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτή την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διάδοσης. Επίσης, ο ρόλος των μεσαζόντων είναι ύψης της σημασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για σύνδεσμο μεταξύ νόμιμου και παρανόμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν το επίπεδο της μεσητείας αυτό, αυτής και να την ελέγξουν, καθώς και να προβούν σε κυρώσεις. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η καταπολέμηση της διάδοσης θα πρέπει να ενισχύσει το, το προληπτικό σκέλος, έτσι ώστε να δράσουμε συντονισμένα ως προς το εμπόριο ε, όπλων, έτσι ώστε να μην να αναχαιτιστεί μάλλον η παράνομη διάδοση. Έτσι θα πρέπει να άρουμε τους κινδύνους μέσα στα πλαίσια της διάδοσης των ε, ελαφρών όπλων, ιδιαίτερα στις ε, υποσύραξη χώρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και ε, να μας πούν γιατί ε, και να τους ευχαριστήσω για ε, τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασαν αυτό το σοβαρό θέμα ε, και το μήνυμα που εξέπεμψαν διότι η πρώτη μου εντύπωση είναι και μπορείτε να με διορθώσετε αλλά μέχρι πριν από δέκα χρόνια Υπήρχαν 600.000 ε, μικρά όπλα σε κυκλοφορία και τώρα οι υπολογισμοί αναφέρονται σε 900.000 πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπήρχε μια, υπήρξε μια αρνητική πρόοδος αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι. Χαιρετήσω λοιπόν την ε, θετική προσέγγιση του τελευταίου ομιλητή του κυρίου Πουατβά διότι αυτό το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη είναι έτσι μια επικοδομητική στάση και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και προβήκατε σε διαφοροποιήσεις μεταξύ της νομίμου και παρανόμου διακίνησης 2 δισεκατομμύρια ευρώ εξάγονται ετησίως σε οπλισμούς από τα κράτη-μέλη και αυτό πρέπει να μας οδηγήσει να σκεφτούμε εάν Χρειαζόμαστε μία συντονισμένη αντιμετώπιση, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με τρίτες χώρες. Να ισχύσουν δηλαδή οι ίδιοι ε, νόμοι για την παράνομη διακίνηση. Αλλά η κυρία Κοπά έχει πρώτο λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. θέλω να ευχαριστήσω θα χρειαστεί κάποια στιγμή να φύγω γι' αυτό αν δεν ακούσω τις απαντήσεις θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις και ελπίζω ότι θα απαντήσετε πριν χρειαστεί να φύγω. Ξέρουμε ότι οι παράνομες αγορές ξεκινούν σαν ένομη διακίνηση. Πώς μπορεί λοιπόν να οδηγήσει, να αποφύγει κανείς την παρέκκληση από μία επίσημη αγορά σε μία παράνομη. Δεύτερη ερώτηση. Ε, πόσο θα επηρεάσει η διακίνηση παρανόμων οπλισμών τους διαμαχόμενους και, ε, σε και πρακτικά πώς εμπινεύεται αυτό σχετικά με τα συμβατικά όπλα. Ξέρουμε ότι όλο και περισσότερο τα κράτη δεν αναφέρουν πόσο διακινούν και εμπορεύονται ε, μικρά όπλα. Είσαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αδιαφάνεια και μία σωστή παρακολούθηση θα μπορούσαμε να βασιστούμε στα προηγούμενα αποτελέσματα μέσω της καλύτερης κοινή παρακολούθησης σε περιφερειακό επίπεδο και πώς όλα αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διακίνηση όπλων. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Η κυρία Γκόμες. Θα πολύ σύντομη για να είμαι βέβαιη ότι θα απαντήσετε στην κυρία Κοπά αλλά θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την ενημέρωση του που βρισκόμαστε και διαβάζοντας αυτά που είπατε και εγώ ανησυχώ γιατί όπως είπε και ο πρόεδρός μας Έχουμε οπισθοδρομήσει από πλευράς ε, ε, αυξήσεως και παρόλα τα μέσα που διαθέτουμε δεν είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στην εφαρμογή ε, σχετικά με τον κώδικα συμπεριφοράς των εξαγωγών. Νομίζω ότι θα ήταν μία σύσταση Ε, για τον κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές των όπλων και για τη στρατηγική κατά της επεκτάσεως της διακίνησης αυτών των μικρών οπλισμών. Από ό,τι θυμάμαι, και ίσως αυτό χρειάζεται μία πλήρη ε, εξέταση το, της μεθοδολογίας την οποία εφαρμόζουν ορισμένα κράτη-μέλη και όχι υποχρεωτικά αυτοί ε, που έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσει όπως η Ιταλία αλλά και άλλες διότι το 2008 διαπίστωσα όταν δεν είχε, ήταν ακόμη δεσμευτικά, ε, δεσμευτικός νομικά ο κώδικας συμπεριφοράς αλλά είχε ήδη θεσπιστεί και προωθούσαμε την εφαρμογή του αντελήφθηκα ότι η χώρα μου είχε ήταν δικτυωμένη ε, και εξήγαγε ε, όπλα αντίθετα προς τον κώδικα συμπεριφοράς τον οποίο είχαν ακυρώσει ε, και επιπλέον υπήρχε και μια τελείως παράνομη οργάνωση της αστυνομίας η οποία τελικά καταδικάστηκε και φυλακίστηκε αλλά δεν ήταν μια καταφανής περίπτωση όπως είπε ο κύριος Μπρόμλεϊ ότι η δίωξη αυτών των παρανόμων ή νομίμων μεσητών είναι κάτι και μεσαζόντων είναι κάτι απαραίτητο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να ελέγχουμε πραγματικά την εφαρμογή ε, αυτών των μέσων διότι ε, ιδάλλως ή δεν θα υπάρχει ε, χρήση είτε θα υπάρχει κατάχρηση των δυνατοτήτων. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε τι αντιφάσεις διαπιστώνεται μεταξύ αφενός της εφαρμογής του πρόγραμμα δράσης του ΟΗΕ και δεύτερον προωθήσεως του ATT διότι θυμάμαι ότι προετών υπήρχε μία πλήρης αντίφαση μεταξύ αυτών των δύο τεχνικών όρων έχει επιληθεί, πώς εσείς αξιολογείτε και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τον στόχο που έχετε καταρτήσει χωρίς να είναι αντιπαραγωγικός. Τέλος, θέλω να ρωτήσω και συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει πολύ περισσότερο τα κράτη-μέλη και να ελέγξουν την νόμιμη και την παράνομη διακίνηση όπλων διότι κάποια εποχή η Επιτροπή είχε κάνει καλή δουλειά με την κυρία Ντανιέλα Ντικοράντο αλλά δεν νομίζω ότι έκτοτε έχει γίνει οτιδήποτε. Υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέληξαν στα δικαστήρια και ίσως ε, θα ήθελα να μου πει η κυρία Γκάντσλαντ Πού βρισκόμαστε με το θέμα αυτής της ενέργειας που έπρεπε να έχει επιληθεί κατόπιν της αποφάσεως του δικαστηρίου για την στήριξη των δυνατοτήτων σε χώρες και περιοχές όπως η Αφρική, η Δυτική Αφρική που προσπαθούμε να περιορίσουμε την ροή όπλων διότι βλέπουμε ότι πρόκειται για όπλα μαζικής καταστροφής. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να μιλήσει. Αν όχι, θα ζητήσω από τους εμπειρογνώμονες να σχολιάσουν. να αναφερθώ σε κάποια από τα ζητήματα που εφήγησαν. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο, ε, το ATT και τη σχέση με το πρόγραμμα δράσης. Θα ζητηθεί ενδεχομένα αργότερα αυτό το θέμα της συνθήκης ε, για το εμπόριο άπλων. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, δεν απαιτείται μόνο το φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό αφορά και τις ε, σχέσεις μεταξύ κρατών και ε, τις αγοραπολισίες. Θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε αυτό το ζήτημα που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη περί εμπορίου όπλων του ΟΗΕ. Μιλάμε για όπλα μαζικής καταστροφής, μέτρα που λαμβάνονται μετά από τη λήξη των εχθροπραξιών και για κανονισμού που θα πρέπει να διεύουν τους κατασκευαστέ. Υπάρχουν μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν και μετά. Επίσης υπάρχουν και κάποια σημαντικά διδάγματα τα οποία θα πρέπει να συναγάγουμε από τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ATT. Υπάρχει έλλειψη σαφών σημείων αναφοράς και Ίσως ε, δεν θα πρέπει να... Μάλλον θα πρέπει να πούμε ότι η ATT δεν έχει κάποιους μηχανισμούς παρακολούθησης ε. Υπάρχει μια γραμματεία η οποία θα πρέπει να συσταθεί. Ένα νομικά δεσμευτικό μέσο θα πρέπει να έχει τέτοιου είδου διευκολύνσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποδυναμώσουμε την πτυχή των, του ελαφρύ οπλισμού στο πλαίσιο της ATT. Να πω κάτι επίσης για το θέμα των πυρομαχικών τον εντοπισμό τους σε εμπόλεμες περιοχές. Υπάρχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα στην Ανατολική Αφρική ιδιαίτερα για να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε την διακίνηση των πυρομαχικών και πώς γίνεται η προμήθεια αυτών. Πρέπει να τονίσουμε ότι περίπου το ίμιση του εμπορίου ανέφερα 8 δις δολάρια αφορούν ε, ένα σημαντικό ποσοστό αφορά τα πυρομαχικά διότι δίχως αυτά τα φορητά όπλα και ολοκλήρης οπλισμός ε, δεν χρησιμεύει θα, είναι, θα λέγαμε σαν νεροπίστολα γι' αυτό λοιπόν επικεντρώνοντας την προσοχή μας ε, στην προμήθεια των πυρομαχικών μας ε, οδηγεί πιο κοντά στο παράνομο εμπόριο. Τουλάχιστον στην Ανατολική Αφρική μπορέσαμε να εντοπίσουμε τρόπους ε, για την παρακολούθηση αυτής της, αυτού του εμπορίου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ε, υπάρχει αυτή η παρακολούθηση, τότε οι χρήστες ε, είναι πολύ πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την χρησιμοποίηση αυτών των πυρομαχικών. Τα πυρομαχικά μπορούν να εντοπιστούν με τον ίδιο τρόπο με, όπως εντοπίζονται και τα όπλα, ο οπλισμός ένοπλες δυνάμεις, ε, οι δυνάμει δυνάμεις ε, συνέβαλαν ε, σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια. Και η διαρροή, θα λέγαμε, αυτών των πυρομαχικών μπορεί να εντοπιστεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εντοπίζονται και τα όπλα. Κάτι ακόμα πρέπει να το εξετάσουμε το ζήτημα ως μια αλυσίδα, δηλαδή πυρομαχικά, όπλα, διακίνηση. Υπάρχουν πολλά σημεία από τα οποία μπορούν να γίνουν διαρροές και να εκτραπεί το εμπόριο από τον νόμιμο στο παράνομο. Έχουμε κάνει κάποιες πρόοδους πάνω σε αυτό. Δεν έχουμε όμως σαφή ιδέα σχετικά με το πιο σημείο της αλυσίδας, ο πιο κρίκος είναι ο πιο αδύναμος. Ξέρετε ότι το να συλλάβει κανείς μια διαρροή σε ένα σωλήνα δεν σημαίνει ότι έκλεισε το, το όλο σύστημα των διαρροών, διότι κλείνει σε ένα σημείο, ανοίγει σε ένα άλλο. σε πολλές περιπτώσεις ε, βλέπουμε ότι έχουν κυκλοφορούν πλαστά πιστοποιητικά, πλαστές αδειοδοτήσεις. Ε, είμαι σίγουρος πως οι συνάδελφοί μου θα έχουν να προσθέσουν κάτι σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Just, I mean, προς το πού υπάρχει διαρροή. Από ό,τι βλέπω από τις έρευνες για τα μικρά όπλα, τα ελαφρά όπλα, για να δούμε πώς ε, γίνεται μέσα στα πλαίσια της ε, φορτωτικής ή μετά τη φορτωτική, νομίζω ότι στο Σουδάν, στο Τσάντ, στην Κεντροαφρικανική ε, Δημοκρατία η διαρροή γίνεται μετά τη φόρτωση και γι' αυτό θα πρέπει να σταθούμε στην ε, κρατική πολιτική γιατί τα όπλα αυτά χορηγούνται σε ε, επαναστατικές δυνάμεις των χωρών αυτών. Μέσα στα πλαίσια της ε, φορτωτικής καθεαυτής οι πολιτικές μας είναι συγκεκριμένες. Μίλησα για τον μηχανισμό εποπτείας για να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση που γίνονται πραγματικά μεταφορές ή όχι ή αποτρέπονται. Έγινε μνήα και στην καταστροφή αυτού του οπλοστασίου. Αλλά αν η κυβέρνηση αργότερα πάρει μια απόφαση, δηλαδή να χορηγήσει αυτά τα όπλα σε επαναστατικές δυνάμεις, το ζήτημα καθιστάται ακόμα δύσκολο σε σχέση με το, όταν, τον έλεγχο για το ποιοι δέκτες είναι νόμιμοι. Το θέμα των μητρώων, του Μητρώου των Ηνωμένων Εθνών, όπως ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι είχαμε αυξανόμενο αριθμό, δηλαδή η αδειοδότηση ζητείται όλο ένα και περισσότερο και ιδιαίτερα από χώρες από τη Νότιο Αμερική όπου υπήρχε μεγάλη περιφερειακή δραστηριότητα. Κάτι το οποίο ενισχύει αυτό το μητρό των Ηνωμένων Εθνών. Ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει πώς γίνεται αυτή η μεταφορά βεβαίως. Η διάσκεψη, το σύμφωνο μάλλον εμπορίας όπλων θα πρέπει να ενισχυθεί. Γιατί από τότε που δημιουργήθηκε αυτό το μέσον κατά τη δεκαετία του 90 μετά δεν χρησιμοποιήθηκε και τόσο ευραίος, όμως έχει μία μεγάλη σημασία αυτό το μητρό. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ε, κατασκευή όπλων από τα κράτη-μέλη. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να αποτιμήσουμε την κατάσταση για να δούμε κατά πόσο έχουν συμπεριληφθεί τα μικρά ελαφρά όπλα σε αυτό το μητρό. Χρειάζεται μία πιο στεναρή στάση από τα κράτη-μέλη. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο συμπεριλαμβάνονται και αυτά τα όπλα απόφαση θα πρέπει να είναι πιο γενικευμένη. Ως προς τις εναλλακτικές πηγές διαφάνειας, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τα δεδομένα και πέρα από τη χαρτογράφηση θα χρειαζόμασταν περισσότερα δεδομένα, ιδιαίτερα σε αμφίβολες ε, περιπτώσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα διεθνή πάνελ, να έχουμε καλύτερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των κρατών. Αυτό ακριβώς κάνουμε, αλλά μπορούν να γίνουν και περισσότερα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό το εγχείρημα μπορεί να μην είναι τόσο δαπανηρό. Δεν θα πω περισσότερα. Για να απαντήσω στην ε, πρώτη ερώτηση ως προς τα προληπτικά μέσα, για να μην περνάνε τα όπλα από το νόμιμο στο παράνομο δίκτυο, έχουμε μία σειρά μέσων. Δεν θα επανεφεύρουμε τον ε, ε, τροχό, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια μέσα έχουμε ήδη στη διαθέσή μας. Ως προς τη μεσητεία, ήδη αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα. Ως προς την εξαγωγή όπλων, υπάρχει η υποψία ότι τα κράτη που είναι τακτική εισαγωγής στέλνουν αυτά τα όπλα σε αντάρτικα. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα ευρύτερα. Ως προς την πιστοποίηση και για το πιστοποιητικό παράδοσης για να γίνουν έλεγχοι θα πρέπει να μην έχουμε μόνο μία σωρία εγγραφών. Δεν μιλάμε για φυσικούς ελέγχους στη χώρα παράδοσης, αλλά μιλάμε για επαληθεύσεις και ελέγχους ως προς τη χορήγηση πιστοποιητικών για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση και στη συνέχεια να μην εξάγουμε προς αυτές τις χώρες. Ως προς το, το θέμα των διώξεων, των ενδεχομένων διώξεων, νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο ε, δίωξη των κακών της υπόθεσης, ας το πούμε έτσι, γιατί το πάνελ εμπειρογνωμόνων δεν έχει τέτοια εντολή, μπορεί να διενεργήσει έρευνα και μόνο. Γι' αυτό σε ορισμένες χώρες υπό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο γίνεται παραβίαση του εμπάργου και Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει, να διενεργηθεί έρευνα από τις δικαστικές αρχές έτσι ώστε να, ε, γίνει, να γίνει δίωξη κανονικά με ορισμό δίκης και ως προς τη μεσητεία θα πρέπει να εφαρμοστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Γκάντσλαντ. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα προωθήσουμε τα ε, συμβατικά εργοστάσια. Μία ακόμη ερώτηση δηλαδή. θα ξεκινήσω με το θέμα της ε, ε, αντίφασης μεταξύ ATT και συμβατικής δράσης όπως είπαν ορισμένοι άλλοι ομιλητές προηγουμένως και εμείς θεωρούσαμε ότι η διάσκεψη ε, αναθεώρησης του προγράμματος έπρεπε να δει πώς θα μπορούσαμε να ενισχυθούμε συμπληρωματικά μεταξύ οργανώσεων και μεταξύ των προτεραιοτήτων που θεώρησα ότι μπορούσαν να λειτουργήσουν ήταν ότι έπρεπε να αυξήσουμε τις προσπάθειες για την διαχείριση των αποθεμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για να μην υπάρχει διαφοροποίηση των αδειοδοτήσεων και θα έπρεπε συγχρόνως να υπάρχει έχει παρακολούθηση από την Ίντερπολ. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι ε, συμπληρωματικά και εδώ δεν πρόκειται για έναν ανταγωνισμό σαν αυτόν που αναφέρατε. Επιπλέον, σχετικά με τις αρμοδιότητες και ε, τα προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει προετών ε, σε σύγκριση με το που βρισκόμαστε τώρα νομίζω ότι καλό θα ήταν να πούμε ότι αυτή η περίπτωση του ΕΚΟΒΑΣ από ό,τι κατάλαβα ήταν ότι η κάθε αρμοδιότητα και κάθε δημοσιονομικό μέσο έπρεπε να συνάδει με τη νομική βάση και να χρησιμοποιείται βάσει αυτής ε, σύμφωνα με το, την οριοθέτηση που είχε γίνει αν πρόκειτο ε, για αναπτυξιακές δράσεις όπως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν είναι CFSP όταν ε, ασχολείται περισσότερο με μία δράση ασφαλείας. Θέλω όμως εδώ να αναφερθώ στη συμπληρωματικότητα ποιότητα των ε, προσεγγίσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι πιστεύω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ενώση έχει ένα συγκριτικό προσόν σε σχέση με άλλους ε, δηλαδή υπάρχουν διάφορα εργαλεία και δεν θέλω να υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεταξύ του, ε, της δράσης σταθερότητας και του CFSP ε, και μάλλον να μπορούν να συμπληρωθούν. Στην εισαγωγή μου λοιπόν είπα ότι το, το μέσων σταθερότητος στηρίζεται από την Ίντερπολ ενώ το Συμβούλιο δρά κατά της ισορρεύσεως στην περιοχή του ΟΑΣΕ και όλα αυτά συνδυάζονται για να καταπολεμήσουν και να καταλήξουν στον ίδιο στόχο με διαφορετικά εργαλεία. Όσον αφορά την αναφορά του που βρισκόμαστε τώρα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην εξαμηνία έκθεση που καταρτίζουμε για την εφαρμογή της στρατηγικής και η έκθεση αυτή είναι αρκετά διεξοδική Δηλαδή προσπαθούμε να ερευνήσουμε ό,τι έχει γίνει, να το δημοσιεύσουμε, να υπάρχει μία ενημέρωση σχετικά με το πού βρισκόμαστε και το ίδιο γίνεται και σχετικά με τη στρατηγική. Μετά, μου ε, ρωτήσατε τι γίνεται με την, ε, τις ε, διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την παραγωγή μικρών οπλισμών με μικρού κόστου στην Ανατολική και ανατολική Ευρώπη που είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ κρατών μελών στα αρμόδιες, στους αρμόδιους οργανισμούς. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον δεν υπάρχουν σχόλια. Uh-huh. So, their suggestion to, to wait. Ε, λοιπόν, προτείνεται να κάνουμε ενό λεπτού διακοπή μέχρι να έρθει ο επόμενος ομιλητής. Τι είναι η επόμενη ομιλήτρια η οποία ήταν εδώ και δεν τη βρίσκουμε. in Προτού όμως ε, ε, προχωρήσουμε σε αυτά θα ασχοληθούμε με την εφαρμογή και την εκμετάλλευση των συστημάτων ε, πλοήγησης δοδηφορικής στην Ευρώπη και τον λόγο έχει ο ομιλητής. Σας ευχαριστώ αναφέρομαι στους, στους ε, ε, σκιώδεις εισηγητές. Ε, θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί είχαμε μία καλή συνεργασία και όπως είπα και στην αρχή ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις πτυχές αυτές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τρόπον ώστε να βρούμε κάποιο τρόπο και να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφαλίσει τη στρατηγική ανεξαρτησία μέσω του συστήματος Γαλιλαίο και ε, στις συζητήσεις μεταξύ ε, σκιωδών διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Γαλιλαίου θα πρέπει να ενισχυθεί και από αυτό το σημείο και πέρα ε, έκανα ορισμένες ε, τροπολογίες ε, και και τονίσαμε, το, τόνισα τα διορυφορικά συστήματα συγχρόνως αναφέροντας πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συστήματα όπου θα έπρεπε να πούμε ότι υπάρχει μία διτή φύση αυτών των μορφών και όσον αφορά τις τροπολογίες έχω τονίσει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει το σύστημα και θα δώσω εδώ συγκεκριμένα παραδείγματα που παρατίθενται ή στις τροπολογίες και που αναφέρονται στην προστιθέμενη αξία αυτών των, των, των συστημάτων. Προσπάθησα επίσης να εξηγήσω ποιο είναι το στρατηγικό ενδιαφέρον αυτού του συστήματος για την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η οποία μπορεί να ενισχυθεί και η ανεξαρτησία αυτή είναι ένα θέμα κλειδί για την άμυνα διότι σε περίοδο κρίσεως οι κίνδυνοι ε, είναι υυξημένοι και ε, ε, είμαστε εκτεθειμένοι στο κλείσιμο των παρόχων οι οποίοι είναι εξωτερικοί ε, προμηθευτές. Γι' αυτό και είναι βασικό να είμαστε προστατευμένοι. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και αναφέρονται στην ασφάλεια του συστήματος. Πρέπει να τονιστεί το θέμα της ασφαλείας και δεν θα έπρεπε τα ε, στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα να ε, μην είναι συνδεδεμένα ή να ερμηνεύονται ε, χαλαρά. Θα πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη βοήθεια και αντιμετώπιση όταν συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες. Ε, με τους κοιόδης εισηγητές καταλήξαμε σε ορισμένες συμβιβαστικές λύσεις διότι θέλαμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το σύστημα και την ε, προώθηση ε, του θέματος ε, ζητώντας να υπάρξει μία αξιολόγηση το 2015. Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστούμε. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία και συγχρόνως αυτό θα μας δείξει μέχρι ποιου σημείου το σύστημα αυτό μπορεί να ελεγχθεί με τον καλύτερο καλύτερο δυνατόν τρόπο εφόσον είναι ένα σύστημα που μας απασχολεί πολύ. Και ε, ε, συμπεραίνω. Η τροπολογία 10 τονίζει ότι ε, είναι βασικό εμπειρογνώμονες αμήνης και ε, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν στην αξιολόγηση αυτού του δορυφορικού συστήματος και ε, εν ανάγκη θα πρέπει να μπορούν επίσης να συμβουλεύσουν την Επιτροπή που θα εποπτεύει το σύστημα αυτό. Ε, τώρα περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και των σχεδόν εισηγητών. Thank Thank you. We have not so many draft persons, but fortunately we have Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι δέχτηκε το αίτημά μου για την ενδιάμεση αποτίμηση, τροπολογία 9, έτσι ώστε να ελέγξουμε την εξέλιξη του προγράμματος. Γενικά αυτή η γνωμοδότηση συμβαδίζει με τις συζητήσεις μας και με την πρώτη συνάντηση των ε, σκιωδών και εγώ θα το διοτύπωνα κάπως διαφορετικά. Θα πρέπει να δούμε τα προγράμματα Γαλιλαίο και Έγνος έτσι ώστε να είναι αυτοδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε καιρό κρίσης. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να αμελήσουμε την πραγματικότητα. Ε, ζούμε σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο, γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε την συνεργασία και την ε, διαλειτουργικότητα. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι ε, ένας δορυφόρος Σογιούς έφερε τον Γαλιλαίο στο διάστημα. Και αυτό δείχνει ότι τώρα μπορούμε να έχουμε ένα μέσο συνεργασίας μετά τον ψυχρό πόλεμο. Η σημασία του Γκαλιλαίου είναι αναμφισβήτητη. Νομίζω όμως ότι η διαχείριση του προγράμματος θα πρέπει να παραμείνει σε χέρια, στα χέρια μιας πολιτικής αρχής και νομίζω ότι όταν υπάρχουν λόγοι άμυνας ή ασφάλειας, τότε θα υπάρχει εξαίρεση, έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με το διεθνές δίκαιο. Όταν μιλάμε για συνεργασία με τρίτες χώρες, δέχομαι τις ανησυχίες που ορίζονται από τις τροπολογίες 4, 7 και 8, αλλά η ουσία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία και αυτοδυναμία έτσι ώστε σε περίπτωση κρίσης να μην χρησιμοποιηθεί το σύστημα κατά ημών όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 25 του σχεδίου κανονισμού. Η ευθύνη αφορά και τη λειτουργία του συστήματος και την ευρύτερη σημασία του. Θα πρέπει να μιλήσουμε για κοινή ε, δράση 552 του κάθετο, κάθετος του 2004, έτσι ώστε η κοινή αυτή η δράση να ενημερωθεί και βλέπουμε ότι προωθείται αναδιατύπωση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάτι για μια πραγματική πολιτική για το σχέδιο Γαλιλαίο που να μπορεί να εφαρμοστεί σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και να ορίσει κατευθυντήριες γραμμές για αποσόβηση μίζωνων κινδύνων. Θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη της Κομισιόν. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα, πώς ορίζεται η αλυσίδα ασφαλείας και πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε, αν χρειαστεί. Ο κύριος Κέλαμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο για αυτή την πολύ καλά προετοιμασμένη γνωμοδότηση. Ένα καθαρά διαδικαστικό, γιατί από όσο γνωρίζω η Ήτρε δεν έχει αποφανθεί και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια γνωμοδότηση. Θα ήταν σοφό, θα ήταν συνετό να προετοιμάσουμε μια γνωμοδότηση όταν δεν ξέρουμε την ουσία της έκθεσης, πώς θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Ως προς τις τροπολογίες και επί της ουσίας, νομίζω ότι οι περισσότερες ε, τροπολογίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ραδιοπλοήγησης. Οι τροπολογίες 2, 4, 5 και 6 αναφέρονται σε θέματα ασφαλείας και είναι πολύ σκόπιμη αυτή η μνήα. Στις προηγούμενες ε, εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας ζητήσαμε τον ορισμό του εθνικού συμφέροντος γιατί μιλάμε για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Σε ορισμένους τομείς ε, νομίζω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένες. Ίσως θα πρέπει να σταθούμε στη σημασία του εθνικ, της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής που έχει μεγάλη σημασία και να μιλήσουμε για την ικανότητα ανάπτυξης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία του συστήματος. Ως προς την τροπολογία 7 εδώ μιλάμε για ενδεχόμενους κινδύνους από τρίτες χώρες. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, συμφωνίες και νομικά μέσα, αλλά θα πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει δράση έτσι ώστε να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία GNSS, η υπηρεσία ραδιοπλοήγησης από τρομοκράτες. Και η τροπολογία 3 μιλά για την ανεξαρτησία της Ένωσης. θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τη χρήση της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής για την ευρύτερη χρήση αυτού του φορέ. Δυστυχώς δεν έχουμε εκπρόσωπο της Κομισιόν. Άρα κύριε Τέρχο θα μπορούσατε εσείς να απαντήσετε στα όσα ακούστηκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα, αν και πρόκειται για ένα θέμα διτού σκοπού, διτής χρήσης. Εδώ όμως αυτό που μας αφορά είναι η μη στερεολογική χρήση. Εξάλλου είναι και η ιδέα η οποία υπερίσχυσε ευθύ εξ αρχής. Φυσικά η στρατηγική ανεξαρτησία είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες και είμαι έτοιμο να εξετάσω τους ποικίλου τρόπους συνεργασίας με τρίτες χώρες και με άλλα δορυφορικά συστήματα. Φυσικά η έκθεση της Επιτροπής Ήτρε είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε του συνεγγύς. Θα δούμε πώς προχωρούν οι συζητήσεις ε, στην ε, Επιτροπή Ήτρε και χρειάζεται να σκεφτούμε τα κράτη-μέλη. Είμαστε τώρα στη φάση να αναζητήσουμε κάποιες εφαρμογέ, αλλά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις. Ε, θα δούμε κατά πόσο παραμένει ένα μη στρατιωτικό σύστημα το οποίο θα την χάνει διαχείριση από μη στρατιωτικού ή θα υπάρχει και η στρατιωτική πτυχή με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και συμβούλων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν εάν τα κράτη-μέλη θα δράξουν αυτή την ευκαιρία να υπάρχει ένα μη στρατιωτικό σύστημα το οποίο όμω θα έχει και ένα δυναμικό στρατιωτικό. Ευχαριστώ. Thank you. So, if there are no more... Ωραία. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν περαιτέρω σχόλια, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της Μεσσίας Διατάξεως, διαπραγματεύει για τη συνθήκη ΟΗΕ όσον αφορά το εμπόριο όπλων, ATT, κυρία Ιετεμάκια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. 17 ή 70 τροπολογίες κατατέθησαν, 70 μάλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το σχέδιο ψηφίσματος έλαβε τέτοια σημαντική συνεισφορά από επαΐοντες συναδέλφους. Πολλές τροπολογίες βελτιώνουν την ποιότητα του κειμένου. Έχω ξεκινήσει σύνταξη των ε, συμβαστικών τροπολογιών και αύριο στις 10 το πρωί θα έχουμε τη συνάντηση των σκιωδών να κάνω μια παρατήρηση εδώ ότι σκοπός της ε, συνθήκης ATT είναι να, διευθυν, να διευθετήσει και να ρυθμίσει το εμπόριο όπλων. Σύμφωνα με τις προφορίες που έχω λάβει, δεν θα συμπεριληφθεί ένα σύστημα εφαρμογής κυρώσεων στην συνθήκη. Η εφαρμογή θα γίνει σε εθνικό επίπεδο και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στις διάφορες φάσεις υλοποίησης της συνθήκης. Αυτό σημαίνει ότι η αναφορά σε ό,τι φορά την ε, μεταφορά όπλων θα πρέπει να είναι ανοιχτή και διάφανη και οι προφορίες ε, να είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες, ε, στα κοινοβούλια φυσικά, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών και στις οργανώσεις αυτής. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει θέσει πολλές ελπίδες, ιδιαίτερα φιλόδοξη και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, είναι μία, ένα από τα διαπραγματευτικά μέρη στη Νέα Υόρκη. Είναι κρίμα. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει ακόμα, δεν εφαρμόζεται μάλλον πλήρως η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία 67. Είναι κάπως πολύ απόλυτη θα έλεγα. Και τώρα πρόεδρε να σχολιάσω κάποιες από τις τροπολογίες εντάχει. Θέλω να αποφύγω επικαλύψεις και επαναλήψεις στο ψήφισμα. Θα καταψηφίσω τις τροπολογίες που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να επαναλαμβάνουν θέματα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε άλλα σημεία του κειμένου. Μία αναφορά αρκεί. Επίσης θα ήθελα να γίνει μια αναφορά στα συμβατικά όπλα. Μάλλον να μην γίνει αναφορά στα συμβατικά όπλα, διότι θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό. Μακρύς κατάλογοι είναι αντιπαραγωγικοί και δεν είναι πρόθεσή μας αυτή. Αναφέρομαι σε τροπολογίε 35 και 6 αλλά και 9 σε αυτές τις τρεις. Στην παράγραφο 8 ζητάω μάλλον στην 7 αναφέρομαι στην ε, επέκταση των κατηγοριών στο μητρό του ΟΗΕ για τα συμβατικά όπλα το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς στη συνθήκη. Ο λόγος για τον οποίο έχω συμπεριλάβει τα φορητά όπλα για τον ελαφρύ οπλισμό αλλά και τα πυρομαχικά οφείλεται στο ότι αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη. Και αυτό πρόκειψε από τις συζητήσεις στην Νέα Υόρκη. Με τα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη συνθήκη, διότι τα φορητά όπλα και ο ελαφρύς οπλισμός προκαλούν σοβαρές καταστροφές, μόλις το συζητήσαμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα ήταν καλό να συμπεριληφθούν στην συνθήκη. Πρόεδρε, χαίρομαι που η Επιτροπή Ασφάλειας ε, έθεσε το ζήτημα αυτό στη μέσα διάταξή της και επιθυμώ να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις για την άψογη συνεργασία τους και να ευχαριστώ και τις μη κυβερνικές οργανώσεις αλλά και τα ερευνητικά Ινστιτούτα τα οποία συνέβαλαν, εργαστήκαμε ε, μέσα σε κλίμα ανεξαρτησίας. Ε, αυτά είχα να πω και τώρα προσβλέπω σε μια συζήτηση τόσο σήμερα όσο και αύριο με τους ποιόδες Κυρία Γκόμες, ε, σκιώδης εισηγήτρια. Ευχαριστώ την κυρία Γιατεμάκη για την εργασία της που προσπάθησε να συμπεριλάβει και όλες τις προτάσεις, σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι. Άκουσα τα όσα μας είπε. Η συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τους εμπειρογνώμονες για τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ όπλισμό έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συζήτησή μας περί της συνθήκης του ΟΗΕ και θα ήθελα να προτείνω κάποιες αλλαγές ή προσθήκες καλύτερα μετά από αυτά που είπε η κυρία Γιατεμάκη την περασμένη Παρασκευή. Παρασκευή είναι. Σε αυτή την ακρόαση που είχαμε νωρίτερα, Μάλλον με βάση αυτή τη συζήτηση να κάνω κάποια σχόλια στις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Συνεχίζει να μην μ' αρέσει η τροπολογία που αναφέρεται στο ότι η βιομηχανία όπλων συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ε, και παραγωγή ναρκωτικών δημιουργεί θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη σε πολλά σημεία του κόσμου και στις δικές μας τις χώρες. Αλλά αυτό δεν είναι ένα καλό επιχείρημα. Ίσως να υπάρχουν άλλα, καλύτερα επιχειρήματα για την στήριξη αυτού του είδους των ε, κατασκευαστικών εταιριών αυτής της δραστηριότητας. συζητήσαμε το ζήτημα της μετατροπής ε, των εργοστασίων κατασκευής όπλων ε, στα κράτη-μέλη, ειδικά στην ε, Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Και αυτό προς όφελος άλλων δραστηριοτήτων, άλλων παραγωγής, πιο χρήσιμες δραστηριότητες και παραγωγές. Ναι, μπορεί να είναι επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται συχνά, αλλά το να κάνουμε εμεί τέτοια επιχειρήματα νομίζω ότι είναι κάπως παράξενο. Είναι, είναι ασυνεπές από πολιτική σκοπιά. Είναι λάθος. Τώρα, σε ό,τι φορά την συμβαστική πρόταση 2, μετά από τις συζητήσεις που είχαμε νωρίτερα με τους εμπειρογνώμονες, είναι αναφορά στην ε, συνθήκη για τα όπλα, αλλά θα ήταν σημαντικό να διευκρινίσουμε την συμπερίληψη φορητών όπλων και ε, λαυρού όπλισμού, διότι αυτά είναι τα όπλα που είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν. Κατανοώ τις δυσκολίες στην συμβαστική πρόταση 3 αναφορικά με τις κυρώσεις που πρότεινα εξ ονόμα της ομάδας μου. Κατανοώ ότι αυτό μπορεί να αποβεί σε βάρος των στόχων σε τη ATT διότι θα δώσει επιχειρήματα σε αυτούς που δεν επιθυμούν αλλά θα μπορούσαμε ίσως να χτενίσουμε κάπως την γλώσσα εδώ και να μην πούμε ότι είναι κυρώσει για, για τις κυβερνήσεις που δεν εφαρμόζουν την συνθήκη αλλά αφορά στην έννοια της ε, δίωξης ε, προσώπων που εμπλέκονται στην παραβίαση της συνθήκης ε, παράνομο εμπόριο κλπ. Τέλος, στην παράγραφο ή μάλλον το πω αλλιώς. Συμφωνώ με τη χρήση του όρου κίνδυνος risk και όχι substantial risk ε, ουσιαστικός κίνδυνος ε, και την συμβαστική πρόταση 6 να προσθέσουμε την έννοια του ελέγχου των δραστηριοτήτων. Κατά τα άλλα προσβλέπω στην αυριανή συνάντηση. Η κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια ε, για την έκθεσή της. Είναι σημαντικό νομίζω να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα εν ώψη της συνδιάσκεψης που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούλιο. Βέβαια, απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του όλου εγχειρήματο του να εγκριθεί δηλαδή μια διεθνή συνθήκη για τον πόριο όπλων, είναι πρώτον ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας της συνθήκης. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα. Δεύτερον, η κάλυψη όλου του φάσματος των συμβατικών όπλων και όχι μόνο των μικρών και ελαφρών όπλων. Τρίτον, η σύσταση μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής της συμφωνίας. Γιατί αυτό θα έχει ασφαλώς νόημα για να αποφεύγεται η εκτροπή από τη συνθήκη. Και πέμπτον, η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών, ιδιαίτερα των κρατών που έχουν τεράστιες εξαγωγές όπλων πολλά των οποίων είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να επισημάνω βέβαια ότι το να προτείνουμε μαξιμαλιστικές θέσεις και προτάσεις έστω και αν συμφωνούμε επί της ουσίας με αυτές ε, ίσως να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα υπό την έννοια ότι δεν θα αναλάβουν όλες οι χώρες να ε, εγκρίνουν αυτή τη συνθήκη ε, ή θα βρεθούν τρόποι παραβίασής της. Ε, η κυρία εισηγήτρια έχει προβεί σε μια σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών. Θέλω να σημειώσω ότι το ΕΠΠ συμφωνεί με την τροπολογία 1, αλλά δεν είμαστε σύμφωνοι με τη διατύπωση «the overthrow of democratically elected governments». Ίσως θα έπρεπε να διατυπωθεί κάπως αλλιώς. Συμφωνούμε με τη συμβαστική τροπολογία 2, καθώς και την 3, 4 και 6. Τώρα στο, στη συμβιβαστική 5, καλύτερα είναι το περιεχόμενό της να παραμείνει στο κυρίως μέρος του ψηφίσματος και όχι να πάει στα recitals. Ε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η συμβολή μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ε, μπορεί να είναι πολύ σημαντική στη συγκεκριμένη αυτή διεθνή συνθήκη. Ε, γνωρίζουμε ότι η παράνομη εμπορία όπλων φυσικά συνδέεται ε, με την τρομοκρατία, με το εμπόριο ναρκωτικών και με διάφορες άλλες παράνομες έκνομες δραστηριότητες στις οποίες πολλές φορές ίσως εμπλέκονται και αντιπρόσωποι κρατών και αυτό είναι που δημιουργεί τις δυσκολίες. Ωστόσο είναι ένα πρώτο βήμα, νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, που πρέπει να γίνει, όχι μόνο γιατί αυτό κατά κάποιο τρόπο στηρίζει την ύφεση και την ειρήνη, αλλά κυρίως και πρώτα απ' όλα διότι η εμπορία όπλων, όπως είπα και πριν, συνδέεται με τις εξόχως έκνομες δραστηριότητες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και που βέβαια η σημερινή παγκοσμιότητα διευκολύνει πάρα πολύ και θα μπορούσε ένα στοιχειώδης έλεγχος του εμπορίου των οπλικών συστημάτων να επιφέρει ύφεση και σε άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγχαίρω και την εισηγήτρια και πάλι. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Κρόνμπεργκ. <clears throat> Ευχαριστώ. Συμφωνώ με το ότι οι συμβαστικές προτάσεις είναι πολύ καλά διατυπωμένες. Έχω δύο ζητήματα που θα θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με το σχόλιο σχετικά με την ε, δημιουργία δέσμευση απασχόλησης ε, να διαγραφεί αυτό το σχόλιο. Τώρα, συμβαστική 5 νομίζω πως ε, έχει πρόβλημα. Τουλάχιστον το σκεπτικό του ψηφίσματος ε, είναι η, μετα, ε, ο έλεγχος και όχι η διακοπή της διακίνησης. Υπάρχουν άλλα άρθρα στο 51. Προτείνω λοιπόν η τροπολογία 51 να ψηφιστεί ως τροπολογία και όχι ως συμβαστική τροπολογία. Τώρα, για την συμβαστική 4 μπορούμε αενάως να συζητάμε τι είναι πιο ουσιαστικό το risk ή substantial risk. Εγώ προτείνω substantial risk, αλλά ίσως θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση. Τώρα, συμβαστική αξία. Πολλά από τα σχόλιά μας έγιναν δεκτά, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στον τελικό χρήστη και τον έλεγχο. Κάποια σχόλια τώρα για τις υπόλοιπες τροπολογίες ε, την έρευνα και ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το στηρίξουμε. Τώρα το πωλήσει όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τώρα τροπολογία 54. Γιατί πρέπει να είμαστε κατά της ιδέας της αλλαγής ε, των κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσαρμογής σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Νομίζω ότι ένας ε, παγκόσμιος κώδικας ε, θα πρέπει να είναι το δυνατόν εγκύτερα στον ε, ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς και θα είναι πιο απλό να εφαρμοστεί από πλευρά μας τώρα, τροπολογία 64, ε, κοινοβουλευτικός έλεγχος, καλή ιδέα, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και την κοινωνία των πολιτών και το ευρύτερο κοινό. στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφορά υπάρχει ήδη διάλογο με την κοινωνία των πολιτών άπαξ ετησίω. Άρα αυτή η τροπολογία δεν λαμβάνει υπόψη τι τρέχουσες πρακτικές και τέλος να σας ζητήσω να δώσετε σαφή εντολή για την εφαρμογή της ATT κάτι που αναφέρουμε στην τροπολογία 59 και να μπορούν να αναλύουν δεδομένα προκειμένου να εντοπίσουν τις ε, διαφορές ε, και τις ε, παραβάσεις στη συνθήκη. Ευχαριστώ. Άλλος, επιθυμεί να το λόγο. Ίσως, ίσως ο κύριος Ντελαπιάτσα θέλει να πει μερικά λόγια. Θέλετε να μιλήσετε. Ένα θέμα μόνο, ένα σημείο ως προς κάτι που έθιξαν αρκετοί για το κατά πόσο θα πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για το γεγονός ότι η Συμφωνία Εμπορίου Όπλων, η ATT, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κοινή μας θέση. Θα θέλαμε να είναι ιδιαίτερα εύρωστη η ATT. Να υπάρχει δηλαδή μια κοινή θέση όπως ίσχυσε το 2008 στον κώδικα συμπεριφοράς. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα διαβαστεί από, τρίτης, από τρίτες χώρες και υπάρχουν ε, πολλοί από τους αδέσμευτους, από τις αδέσμευτες χώρες που θα ε, πρέπει να δούμε πώς θα ερμηνεύσουν αυτό το πλαίσιο. Γιατί μιλάμε για πολυμέρεια, για πολυμερείς σχέσεις και πολλοί από αυτές, από αυτούς δεν θέλουν να ενισχύσουν το σύστημα μεταφοράς ελέγχου. γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολυμέρεια του συστήματος σε διεθνές επίπεδο. Ο εισηγητής, η εισηγήτρια, με συγχωρείτε, θα ήθελα να σας συγχαρώ όλους. Αύριο στις 10 θα συνεχίσουμε και νομίζω ότι θα φτάσουμε σε πολύ καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν κανείς άλλος δεν θέλει το λόγο, Πιστεύω ότι τελειώσαμε για απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.